Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ξεκινούμε τις εργασίες μας αμέσως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την προσέλευσή σας εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Ως συνήθως να κάνω τις ε, παρατηρήσεις μου. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο Υπάρχει διερμηνία στις γλώσσες των πλήρων μελών της ε, Επιτροπής μας. Θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Εγκρίνεται. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι δύο σημεία της ημερήσιας διάταξής μας θα συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών αμέσως μετά την, ε, το πρώτο θέμα, την ανταλλαγή απόψεων με τον καθηγητή Σβέν Μπίσκοπ. Θα συζητήσουμε δύο θέματα και κλεισμένων των θυρών. Ένα που αφορά την κατάσταση στη Συρία, στο Χαλέπι συγκεκριμένα, και το δεύτερο θέμα που αφορά την κατάσταση γύρω από την ασφάλεια στα Βαλκάνια. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε γκρίνει την ημερήσια διάταξη και πάμε τώρα να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 12 και 13 Οκτωβρίου του 2016. Η προθεσμία υποβολής σχολείων ενστάσεων είναι ε, σήμερα μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας. Ενημερώστε παρακαλώ σε αυτή την περίπτωση αν έχετε δηλαδή παρατηρήσεις. Αν ωστόσο δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ενστάσεις, θεωρούνται, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί και τα πρακτικά. Και τώρα να περάσω αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω την ε, δυνατότητα να ε, υποδεχθούμε εδώ τον ε, κύριο Σβέν Πίσκο που είναι ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γάντης και στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Έγμοντ. Θα έχουμε λοιπόν μια ανταλλαγή ε, απόψεων όσον αφορά την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής και συγκεκριμένα τον αντίκτυπο της παγκόσμιας στρατηγικής στις διατλαντικές σχέσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη σήμερα, οπότε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Μπίσκοπ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ μετά από αρκετό καιρό. Νομίζω από την ε, προηγούμενη θητεία έχω να έρθω του Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι έχει αλλάξει και η σύνθεση της Επιτροπής. Πολύ σύντομα θα σας μιλήσω τον αντίκτυπο της παγκόσμιας στρατηγικής και την εφαρμογή αυτής, γιατί πρέπει να πω ότι δεν βλέπω και πολύ εφαρμογή, άρα και όχι πολύ μεγάλο αντίκτυπο, δυστυχώς μέχρι στιγμή. Ωστόσο, ε, φαντάζομαι ότι θέλετε να σας, ε, να, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Θα χωρίσω τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις σε δύο τμήματα. Ένα που θα αφορά την άμυνα και ένα που θα αφορά ε, την διπλωματία και, το, και τις εμπορικές σχέσεις. Γιατί αυτά τα δύο αλληλοδιαπλέκονται. Όσον αφορά την άμυνα, αν εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει η παγκόσμια στρατηγική, αυτό φυσικά θα αποβεί σε όφελο των διατλαντικών σχέσεων. Γιατί φυσικά η συζήτηση για τον καταμερισμό των βαρών ε, ε, και ε, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τους Αμερικανούς ε, στον τομέα της άμυνας. Αυτό ε, θα αποτελέσει ένα σημαντικό ζήτημα άπαξ και λάβει τα καθήκοντά του ο Ντόναλτ Τραμπ. Ε, το έχει θέσει το ζήτημα αυτό με μεγαλύτερη σαφήνεια από κάθε άλλον προκάτοχο του και το γεγονός ότι έθεσε και το ζήτημα του άρθρου 5 είναι ε, αρκετά ενδιαφέρον. Αλλά το, η συζήτηση αυτή ε, ξεκίνησε πρώτα την περίοδο του, του Kennedy, Δεν είναι καινούργια. Πάντω είμαι πεπισμένο ότι ο μόνος τρόπος ε, να ενισχύσουμε εμεί οι Ευρωπαίοι τι αμυντικές μα προσπάθειε ε, προσπάθειες είναι ε, να αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές δομές. Ειλικρινά όμως δεν βλέπω να υπάρχει πρόοδος παρά τα πολύ λεπτομερή συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου ε, έκανα κάτι ε, ε, μια ζεβολιά έκανα. Γιατί πήγα και ξανακοίταξα τα συμπεράσματα συμβουλίου του Δεκεμβρίου του, του, του 2013. Ε, αν τα συγκρίνεις τα δύο κείμενα, δεν είναι σαφές πότε συνετάχθη το, το καθένα. Κάνουμε δηλαδή κύκλους γύρω από τον εαυτό μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δηλώσει ότι μπορεί να ε, αποτελέσει ένα παράγοντα διευκόλυνσης. Μπορούμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει διευκολυντικά, αλλά ε, ταυτόχρονα δεν είναι έτοιμη ή δεν γνωρίζουμε αν είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στην πράξη αυτές τις, ε, τις Και δεν ξέρουμε αν κάποιος έχει πραγματικά πρόθεση να κάνει το οτιδήποτε. Από την δημοσίευση της στρατηγικής φυσικά ε, συνέβη το Brexit. Υπάρχουν δύο ε, γαλλογερμανικές προτάσεις και γαλλοσπανικές, αλλά ακόμη και αυτά τα κράτη-μέλη δεν έχουν δείξει σημεία ότι πράγματι θέλουν να αναλάβουν δράση σε αυτά τα θέματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, στο Ινστιτούτο είχαμε κάποια στιγμή πρόσφατα μία συνάντηση από την Γερμανία, από το Ινστιτούτο Στρατιωτικών Μελετών. Ε, υπήρξε λοιπόν μια συνάντηση ε, όπου υπόθηκε από τους Γερμανούς ότι η Γερμανία θέλει πραγματικά να αναλάβει δράση. Ήταν πολύ θετικό το κλίμα, υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός. Τέλειωσε η συνεδρίαση, πάω και διαβάζω τα email μου ως συνήθως και μου στέλνει ένας Γερμανός στρατιωτικός φίλος ε, ένα email, ο οποίος είχε ε, μόλις συμμετάσχει συμμετάσχει ε, στην ε, συνδιάσκεψη του Υπουργείου Άμυνα. και τι ήταν το, το ε, μήνυμα που μου έστειλε ήταν ότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες, ε, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία στο δραστηριοτικό τομέα, ε, το, το, το ε, μήνυμα λοιπόν ήταν ε, αντιφα... τα μηνύματα λοιπόν είναι αντιφατικά είναι σαν σκοτσέζι κοντούς μερικές φορές ε, αν συγκρίνει κανείς αυτά που ακούγονται Επίσης δεν υπάρχει ακόμη σαφήνεια για το τι ακριβώς καλούμαστε να κάνουμε γιατί έχουμε αποφύγει τη συζήτηση γύρω από το επίπεδο της φιλοδοξίας που υπάρχει η παγκόσμια στρατηγική είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά την άμυνα. Και είναι λίγο ηρωνία γιατί κατά τη σύνταξη ε, ε πολλοί ε, ε, είχαν εκφράσει την άποψη ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θέτηση είναι αρκετά φιλόδοξη, βάζει καθήκοντα στις, στις ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης, την προστασία, την, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αναφέρει συγκεκριμένα τι, ε, ότι αυτά τα, τα καθήκοντα ε, θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε ακόμη και χωρίς τις ΕΠΑ, αν, ε, αν χρειαστεί. Αυτό φυσικά, αυτά, αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο ε, στρατιωτικής βούλησης για, δράση. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα οι, οι Ευρωπαίοι ε, αναπτύσσουν στρατεύματα και ε, βασίζονται στους Αμερικάνους ε, για, την, για τις στρατιωτικές τους ανάγκες. Αν θέλεις όμως στρατιωτική και επιχειρησιακή αυτονομία δεν μπορείς να βασίζεσαι στους Αμερικάνους. Επιπλέον, τη στιγμή που θα αποχωρήσει η Βρετανία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμβολή της ε, επίσης θα καταργηθεί. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, οι, βρασ... οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν δεν θα... Ε, από το χάρτη. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και αν υπάρχει απειλή για την Ευρώπη αυτή θα είναι απειλή και για τη Βρετανία. Και ε, σε περίπτωση που η Ευρώπη αποφασίσει να αναλάβει δράση, φυσικά ε, αυτό θα αφορά και την Βρετανία. Αλλά η Βρετανία θα είναι εκτός των επίσημων δομών. Άρα, αν θέλει κανείς μια πραγματική παγκόσμια στρατηγική, πρέπει να ε, ε, αναθεωρήσει το επίπεδο φιλοδεξίας. Αλλά τα κράτη-μέλη μέσω του Συμβουλίου αρνήθηκαν ακριβώς να κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν κάνουμε έναν κύκλο. Ε, όσον αφορά τις απαιτήσει ε, ικανοτήτων, το Συμβούλιο ε, έδωσε, υποτίθεται νέα εντολή, αλλά ε, επί της ουσίας δεν υπάρχει συγκεκριμένη εντολή για το πόσες επιχειρήσεις και σε ποια κλίμακα θέλουμε πραγματικά να είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε Κινούμε, λοιπόν, κινούμαστε λοιπόν γύρω από έναν κύκλο. Δηλαδή υπάρχει η παγκόσμια στρατηγική ε, με την ανάγκη ε, αύξησης της, του επίπεδου φιλοδοξίας. Υπάρχουν τα, τα, ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία κινούνται σε, αντίθεση, σε αντίθετη κατεύθυνση και έτσι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, οι στρατιωτικοί να κατανοήσουν ακριβώς πού κινούμαστε. Αν θέλουμε να αναλάβουμε δράση και να γνωρίζουμε για ποιους ε, στόχους ακριβώς ε, θα αναλαμβάνουμε δράση, πρέπει να ορίσουμε τη μεθοδολογία συγκεκριμένα και κατά τη γνώμη μου ε, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα από την αμυντική συνεργασία προς την αμυντική ολοκλήρωση. Τώρα βρισκόμαστε περισσότερο στο στάδιο της αμυντικής συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κάποιες προμήθειες ad hoc από καιρούς καιρών και αναπτύσσουμε και ορισμένε πλατφόρμες κοινέ, αλλά στη συνέχεια αυτά καλούνται να τα υλοποιήσουν εθνικά τμήματα, εθνικές μονάδες, ε, ε αντί ε, ε, να δημιουργούνται δηλαδή πολυεθνικά τμήματα σε μόνιμη βάση. Αυτά είναι κάποια, κάποια, κάποια παραδείγματα. Η γερμανογαλλική συνεργασία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η συνεργασία μεταξύ Βελγίου ε, και ε, κάτω χωρών στον, στο ναυτικό, αλλά αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις ικανότητές μας πρέπει να ε, οικοδομήσουμε πολυεθνικά τμήματα όπου αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από, από, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σκεφτείτε μια βασική ε, μονάδα, μια βασική δομή στην οποία μπορούν να ε, συνεισφέρουν όλα τα κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούν να αξιοποιούν ένα, έναν κοινό πυρήνα πόρων. Αν λοιπόν αποφασιστεί να πάμε σε ένα τέτοιο σε, ένα τέτοιο επίπεδο ε, αμυντικής ολοκλήρωσης ε, χρειάζεται να εξασφαλιστεί ε, ότι ένα, νομικό πλαίσιο που θα είναι δεσμευτικό όσον αφορά τις συνεισφορές των συμμετεχόντων. Δεν χρειάζεται να είναι μόνιμο χαρακτήρα αυτό. Μπορεί να, να επικαιροποιήσει κανείς το, το, το μοντέλο της ε, γερμανική στρατιωτικής συνεργασία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συμμετέχει η, η, Γαλλία βέβαια. Ή μπορεί να δημιουργήσει και κάτι εντελώς καινούριο, αλλά ε, εκεί χρειάζεσαι και ένα νέο ε, νομικό πλαίσιο. Γιατί κατά τη μετάβαση από τη συνεργασία στην ολοκλήρωση μπορεί να, να γίνει μόνο μία φορά η πραγματική ολοκλήρωση, συγχώνευση δηλαδή ε, στρατιωτικών μονάδων. Μπορεί κανείς να, να πάρει ε, την, την ΠΕΣΚΟ, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες Β και Γ του, του εθνικού πλαισίου. Ακούω πολλούς που θεωρούν ότι το ΠΕΣΚΟ ε, είναι στην ουσία επιχειρήσεις των κρατών μελών, δηλαδή το, η Α και η Β χώρα κάνουν το, το πρόγραμμα Χ και οι χώρες ΓΔ Δέλτα κάνουν το, το, πρόγραμμα ε, Ψ. Αν δεν αξιοποιηθεί θα, είναι μια χαμένη ευκαιρία το, ΠΕΣΚΟ. Βλέπω λοιπόν ότι ελπίζω ότι έως το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν ε, ανακοινώσεις και θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα όσον αφορά τις ε, προθέσεις των κρατών μελών. Γιατί αλλιώς το σχέδιο εφαρμογής απλά θα παραμείνει αυτό που ε, λέει, ότι ένα σχέδιο δηλαδή. Δεύτερο κομμάτι των ε, ε, σχολείων μου, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα υπάρχουν εντάσεις με τις ΕΠΑ, είναι η διπλωματία. Μέχρι στιγμής, στην ουσία περιμένουμε. Υπάρχει ένα μοντέλο που επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που αναλαμβάνει μια νέα ε, Αμερικανική κυβέρνηση ακούγονται πολλά, συζητιόνται πολλά και στη συνέχεια απλά περιμένουμε έως ότου ο Τραμπ να κάνει κάποιες, ε, κάποια τηλεφωνήματα, να δει και κάποιους εταίρους του και ε, στη συνέχεια να ανακοινώσει ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Αλλά δεν βλέπω κάποια δραστήρια ε, κίνηση για το ποια είναι η δική μας ε, στάση όσον αφορά τη διπλωματία και μια δική μας πρωτοβουλία να αναλάβουμε επικοινωνία με τις ΗΠΑ. Και ε, περισσότερο ασχολούμαστε με την άμυνα παρά με την ε, διπλωματία. Βλέπω ε, ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας είναι ψηλά στην ατζέντα μας και παρόλα αυτά δεν αναλαμβάνονται δραστήριες κινήσεις. Δεύτερο θέμα, η σχέση μας με το Ιράν για τους Ρεπουμπλικανούς αποτελεί ένα, ένα εμβληματικό θέμα ε, ενδεχομένως ε, θα μπορούσε ακόμη και να ε, καταργηθεί η συμφωνία η οποία πετεύχει για να κάνει και την, μια κίνηση σύμβολο το, το, ο, ο Τραμπ. Αυτό νομίζω ότι δεν επιδέχεται αμφιβολία. Είναι κόντρα και στα οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια συμφωνία. Δυνατόν να έχουμε σταθερότητα στην περιοχή του κόλπου εάν δεν εμπλέκονται οι υπέρ. Δηλαδή τελείω αντιπαρικό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί προς την κυβέρνηση Τραμπ. Επίσης, υπάρχει ο φόβος ότι ο νέος πρόεδρος θα τα βρει με τον Πούτιν. Βέβαια, το ότι θα προσπαθήσει να κλείσει κάποια συμφωνία με την Ρωσία θα προφερθεί ο θετικό, αλλά δεν μπορούμε να ποντάρουμε σε αυτό τόσο πολύ, γιατί νομίζω ότι έφτασε η Ρωσία το σημείο στο οποίο και αυτή έχει συμφέρον να πάψει τον πόλεμο στη Συρία. Να παραμείνει η κυβέρνηση Άσαντ. Ήδη αναπόφευκτα έγινε η επέμβαση εδώ και τόσους μήνες αλλά τώρα η κατάσταση έχει παγώσει, δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει τον πόλεμο ο Άσαντ. Άρα τι νόημα έχει να συνεχίσει τον πόλεμο η Ρωσία. Άρα είναι κοινό το συμφέρον όλων μα, Αμερικανών, Ευρωπαίων, Ρώσων. Α βέβαια ακριβώ γι' αυτό δεν μπορεί κανεί με οποιοδήποτε τίμημα να κάνει συμφωνία με του Ρώσους, Ιδίω με αντάλλαγμα Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία. Όλοι ξέρουμε βέβαια ότι ποτέ θα δώσουν πίσω την ε, Κρυμαία ούτε επίσης ότι θα προσφέρουμε θέσεις στον ΝΑΤΟ στην ε, Ουκρανία. Οπότε υπάρχει συμφωνία του Μίνσκ που θα πρέπει να παραμείνει σεβαστή, δηλαδή πλήρης αποκατάσταση των Ουκρανικών συνόρων. Να σταματήσει αυτή η εξέγερση στην Ανατολική Ουκρανία Και πού να φανταστώ ότι ο Πούτιν μπαίνει στον πειρασμό να κλείσει αυτή τη συμφωνία με τον ε, ε, Τραμπ. έτσι θα αναδεχθεί ως μέγας ηγέτης. Αλλά δεν την άλλη θα κρατήσει και πολύ αυτή η περίοδος χάριτος που έχουν τις άγαστες σχέσεις. Οπότε τελικά μπορεί να του ανοίξει όρεξη αντί να κάνει συμβασμό. Και αν θέλει να κλείσει συμφωνία ο Τραμπ με τη Συρία, πώς θα την κάνει αν δεν εμπλακούν και οι Ιρανοί. Άρα θα πρέπει να διαλέξει ο Τραμπ. Θα κάνει συμφωνία με τη Ρωσία ή θα καλύψει και το Ιράν. Τέλος πάντων, το τελευταίο που θα σας αναφέρω είναι η Ασία. Ήδη ο Ιάπων Πρωθυπουργός πήγε στον ε, πύργο, στο μέγαρο του Τραμπ και έτσι αν έχουμε ένα πολυμερές πλαίσιο ε, στα πλαίσια του ειρηνικού αυτό είναι θετικό για τη σταθερότητα. Αλλά εάν ο Τραμπ καταλήξει το TTIP και δεν κάνει τίποτε άλλο και αρχίσει και προστευτική πολιτική σχέση με την Κίνα, ε, τότε θα υπάρξει ένα κενό στην Ασία. Και η Κίνα τώρα θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα να το κάνει αυτό. Για Ιαπωνία, για Βιετνάμ, που θα πρέπει να μην μπουν στη σφαίρα επιρροής της ε, Κίνας. Θα περιπλακούν τα πράγματα. Και ακόμα χειρότερα για τι Φιλιππίνες που ήδη έχουν προσεγγίσει την Κίνα. Οπότε υπάρχουν και άλλε επιπτώσει. Σε μια τέτοια σφαιρική στρατηγική θέλουμε να επιταχύνουμε το να υπάρξει συμφωνία στην Ασία με Βιετνάμ ιδίως. Η μεγάλη σημασία πολιτική, γεωπολιτική και να είναι εγγύτης ασφάλειας η Αμερική. Αλλά το FTS επίσης είναι ένα του για αυτές τις που θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις από την Κίνα για να το καταφέρουν. Είναι σημαντική η εμπορική μας παρουσία και από πολιτικής πλευράς. Άρα κάθε κίνηση εκεί πρέπει να σκεφτούμε καλά. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα ε, τα οποία νομίζω ότι μπορεί να ασκήσει δυναμική διπλωματία η Ευρώπη, αλλά δεν το διαπιστώνουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο και ούτε αποτελούν αυτά τα θέματα προτεραιότητες της ε, είπα, της εκπροσώπου για την παγκοσμία στρατηγική. Άρα, Είναι πολύ ε, πιθανό να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από τον Τραμπ η Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί και να χαρακτηρίσει μια στρατηγία από νωρί. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ για την εισήγηση που κάνατε και τώρα να δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Γκάλερ πρώτος ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίσχοπ για ε, την παρουσίαση αυτή. Ομολογώ ότι συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό μαζί σας. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση των φιλοδοξιών, το επίπεδο των φιλοδοξιών μας, σωστά είπατε ότι αν κοιτάξουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου 2013 και τα όσα δηλώνονται τώρα. Καλά, το ίδιο κείμενο είναι. Κάνουμε κύκλος, κυνηγάμε την ουρά μας. Βλέπω και για απροθυμία να υλοποιηθούν ε, αυτά που έχουν συζητηθεί, ε, όπως η ΠΕΣΚΟ που είναι η μόνιμη ε, διαρθρωμένη συνεργασία και για την οποία μιλούν όλοι. Εγώ είχα την αίσθηση ε, ότι η Υπουργό Αμήνη τη Γερμανία ε, το υπερασπίζεται στεναρά. Την έχω ακούσει και ο ίδιο να το λέει, ότι θέλουμε τώρα να την ενεργοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία. Και είναι πραγματικά ενοχλητικό όταν λέτε ότι πήγατε στη Βόνη και ακούσατε σε μια διάσκεψη ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ελπίζω κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε δεν αρκεί να το δηλώνει ένα κράτος μέλος. Θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Συμφωνώ επίσης και με την εκτίμησή σας ότι δεν υπάρχει έτσι κάποια πρωτοβουλία απέναντι στη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Να αναλάβουμε εμείς την πρωτοβουλία. Εγώ θα επιθυμούσα Στη παρούσα φάση η κυρία Μογκερίνη να μεταβεί στην Ουάσιγκτον και να βρει ε, την είσοδο του μεγάλου Τραμπ. Τώρα δεν είναι η ώρα να πει η κυρία Μογκερίνη τι θέλουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Και να εξηγήσει και στον κύριο Τραμπ κάποια βασικά μηνύματα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και πολλή ώρα και να ακούσει τι λεπτομέρειες. Γιατί άμα πάνε 28 υπουργοί εκεί θα το ζαλίσουνε. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να λάβουμε εμείς πρωτοβουλία και να πούμε τι περιμένουμε εμείς Ευρωπαίοι και όχι απλώς να πάμε εκεί και να ρωτήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσά. Αυτό το ξέρουμε. Θέλουν περισσότερε στρατιωτικέ δαπάνες. Το 2% στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ζητούν οι Αμερικανοί. Έχει υποφασιστεί ήδη αυτό στο ΝΑΤΟ. Συμφωνώ απολύτω λοιπόν μαζί σας. Δύο ερωτήσει έχω για την δική σας εκτίμηση. Και οι δύο έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση. Πρώτον, δεν αναφερθήκατε ακόμα σε αυτό, αλλά κυκλοφορεί η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Ομιλικού Ταμείου. Και Έχουμε και το μηχανισμό Αθηνά ε, για ε, τις αποστολές της ΕΠΑ, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας. Αλλά αυτά είναι κυρίως στα χέρια των κρατών μελών τα οικονομικά που συμμετέχουν με τις γνωστές συνέπειες. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν καθόλου ή πολύ περιορισμένα γιατί δεν μπορούν ας πούμε, να στέλνουν και το ναυτικό τους γιατί θα υπομισθούν όλο το κόστος. Οπότε, ερωτώ, πώς εκτιμάτε την προθυμία αυτός ο μηχανισμός Αθήνα να Ατένα να επαναδιαμορφωθεί έτσι ώστε να χρηματοδοτείται από έναν άλλον κοινό κορβανά των κρατών μελών, ένα ταμείο για την άμυνα. Και από την άλλη, τι πιστεύετε για την ιδέα που ακούγεται να προχωρήσουμε σε κοινά προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Μηδικό Ταμείο, European Defense Fund. Και από τη δική μου τη χώρα έχω ακούσει θετικές αντιδράσεις. Με τους γνωστούς όρους και προϋποθέσεις. Αλλά αν κάναμε κάτι από κοινού, μπορεί να υποστηρίζαμε και κοινά έργα και θα ήταν και πιο φτηνές ενδεχομένως κάποιες προμήθειες με ε, αυτή την οικονομία κλίμακας, με συγκεκριμένο συνδυασμό και δημόσιες προμήθειες. Δυναμικό υπάρχει. Πολιτική βούληση υπάρχει, κατά τη γνώμη σας. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστούμε, κύριε Φρόιντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Μπίσκοπ, και συμπάθαμε που άργησα λίγο Αλλά τα περισσότερα πόσα είπατε τα άκουσα. Δεν ξέρω είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων τέλος πάντων πριν τα Χριστούγεννα γιατί ε, αυτή τη φορά περίεργο συμφωνώ με τα περισσότερα από ο κύριος Γκάλερ. Από την αρχή ήμουνα υπέρ του να έχουμε μια ενεργή, μια δυναμική εξωτερική πολιτική στην Ευρώπη. Όπως είπε και ο Μίχελ. Επιδραστική, ε, αποφασιστική. Ανέκαθεν το λέγω αυτό. Α, να πάει η Φεντερίκα Μαγκερίνη στον ε, Τραμπ. Εντάξει, όσο και αν έχω τι επιφυλάξει μου, και από το 98 παγκόσμια από κοντά τις ε, αμερικανικές εκλογές και ποτέ, ποτέ δεν σε τόση απογοητευσή όσο φέτος. Με την νέα κυβέρνηση, με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο, γιατί δεν έχεις από να τον πιάσεις, από πού να, να, τον καταλάβεις εκτός από αυτή την ε, προκλογική εκστρατεία. Και με αυτά που έλεγε, πού να βρούμε ακτίνα αισιοδοξία να έχουμε. Τέλος πάντων, διάβασα στο Bloomberg τη προάλλε που έλεγε ποιο είναι ο οδηγός του απεσιόδοξου για το 2017. Το κάνανε αυτό και για το 2016 και πέσανε μέσα για τον Τραπ πέσανε μέσα και για τον Brexit. Βέβαια πέσανε έξω για άλλα τα οποία δεν τα τονίζουν. Αλλά να σας πω που τα πήγαν καλά ή τέλος πάντων αυτά που περιμένω ότι θα πέσουν μέσα. Ότι ο Πούτιν θα σταματήσει τους ε, χάγες που κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις. Δεν θα υπάρχει ανάμειξη στα αμερικανικά πράγματα. Η Μέρκελ θα αναγνωρίσει τα όσα κάνουν σε Συρία και Ουκρανία οι Ρώσοι. Η Κίνα ξεκινά οικονομικό πόλεμο. Ε, αυτό βέβαια πώς να το αποκλείσει κανείς. Εκείνο θα κάνει ρεκόρ ύφεση, η Βόρεια Κορέα είναι πρόβλημα για τόσο καιρό και όμως τελικά καταφέρνει να εγκαταστήσει τα πυρηνικά να έχει ένα πύραυλο μπορεί να χτυπήσει τις ΕΠΑ Η Λεπέν ε, κερδίζει σε εκλογέ. Πολλά, πολλά λένε ότι θα γίνει. Για τα δύο τελευταία, εγώ δεν νομίζω ότι, ότι θα, θα χάσει εκλογέ. Η Μέρκελ ότι θα κερδίσει η Λεπέν. Αλλά δεν ξέρω. Θέλετε να σχολιάσετε τον κατάλογο από αυτά τα θέματα, αυτέ τις προβλέψεις και θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά πιο δυναμικά και να ακούει τη φωνή της ενιαία. Περισσότερο από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριος Γιούρεκ. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za... Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και εγώ το καθηγητή κύριο Πίσχοπ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ δε περισσότερο που οι εμπειρογνώμονες πάντα είναι πιο ελεύθεροι στο λόγο τους και μπορούν να λένε πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα και σαφή, πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς. Θέλω να σας ερωτήσω λοιπόν το εξής κύριε καθηγητά. Ποια είναι τα προβλήματα ασφαλείας ε, που μπορεί να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των ε, μελών της. Τι εννοώ. Στην πολιτική ασφαλείας δεν ταυτίζονται πάντα τα συμφέροντα. Ε, Διεθνώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει μεγάλο κύρου, συμμετέχει στην επίλυση μεγάλων ε, διεθνών προβλημάτων όπως είναι η σύραξη στη Συρία ε, που είναι, δεν είναι μόνο πόλεμο εκεί, είναι και ανθρωπιστική καταστροφή και ένα πρόβλημα που απειλεί την ίδια την ασφάλεια της Ευρώπης. Επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ λόγω και των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τον πόλεμο και αυξάνονται. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία ε, διετία, ε, δεν κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Ασχολούμαστε με τους πρόσφυγες, αλλά δεν ασχολούμαστε με την προσφυγική κρίση για να αντιμετωπίσουμε ε, την αιτία της κρίσης. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με το σημαντικότερο πρόβλημα που είναι η ασφάλεια των ίδιων των κρατών μελών της. Δηλαδή, η πολιτική ασφαλεία είναι κάτι που ε, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάθε κράτος ξεχωριστά. Οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να βγουν και να πούν το κράτος είμαι εγώ και αυτό που με ενδιαφέρει μόνο είναι η ίδια μου η χώρα και ο λαός μου. Είπατε ότι η Κρυμαία αποκλείεται να επιστρέψει στην Ουκρανία. Πολλοί πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πιστεύουν αυτό. Άλλο είναι αν το λένε κιόλα. Δεν το ξεστομίζουν. Αλλά άλλο είναι να το ξέρεις και άλλο είναι να λες ότι δεν θα κάνω τίποτα. Ούτε στο ΝΑΤΟ. Για να διαφυλάξουμε την ε, δαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένης και της Κρυμαίας. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα όμως εκτός από όλα αυτά η πρόεδρός μας χτες διοργάνωσε μια δημόσια ακρόαση με τα τάρους της Κρυμαίας, τον Μουσταφά Τζεμίλε και άλλους. Έγινε μια συνάντηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε πολιτική διαδήλωση, όχι εκδήλωση μόνο. δεν έχουμε καταλάβει ότι το ένα έβδομο του πληθυσμού της Κρυμαίας είναι αυτόχθονες ηθαγενείς, τατάρι. τατάρι. Και είναι και βαρόμετρο της ε, εξέλιξης της κοινωνίας. Η Ρωσία είναι κατευθυνόμενη δημοκρατία. Είναι ένα είδος επίφασης δημοκρατίας. Γι' αυτό μπορεί και να κατευθύνεται ή να χειραγωγείται. Γιατί η ηγεσία διατηρείται στην εξουσία υπογραμμίζοντας αυτό τον ηγετικό χαρακτήρα και ρόλο που έχει. Ε, η Πρόεδρος ασχολείται με την Κρυμαία, ε, παρακολουθούμε την Κρυμαία, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε απαθείς θεατές ή τα κράτη που είναι τα πιο ενδιαφερόμενα, τα πιο κοντινά να δηλώνουν και να δείχνουν το ενδιαφέρον τους, θα πρέπει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δραστηριοποιείται. Επόμενη ερώτηση. Η συμφωνία με τη Ρωσία, είπατε, η συνεννόηση. Εγώ πώς το βλέπω. Για τη Συρία προφανώς ε, πρόκειται, αλλά τίθεται και το θέμα τι, πώς να συνεννοηθείς με τη Ρωσία το 1 τέταρτο των κρατών μελών που συνορεύουμε την Ουκρανία ή και με τη Ρωσία ε, περιμένουν από εμά να δραστηριοποιηθούμε. Η πολιτική του κυρίου Πούτιν είναι σκέτη προπαγάνδα. Και στην εξωτερική πολιτική προσπαθούμε έτσι κάπως να κάνουμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε τον Πούτιν, έτσι κάπως ελαφρά και συγκρατημένα, δεν είναι πολιτική ισορροπιών. Όταν κάνει κάποια βήματα η Ρωσία, κάνουμε εμείς ε, ε, κάποια άλλα βήματα για να επανέλθει η ισορροπία. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο χλιαρά. Και Υπάρχουν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφυλακτικά εξ αυτού του λόγου. Δεν μιλώ για τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ε, είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά μιλώ για την ενιαία δράση. Και θα πρέπει να προβληματιστούμε. Τι θέλουμε τελικά, τι μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να έχουμε παρουσία στη διεθνή πολιτική σκηνή. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, θέλουμε να τονίσουμε, να αυξήσουμε το γόητρο και το κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως το κάθε κράτος μέλος έχει τα δικά του συμφέροντα. Και η Ένωση είναι ένα άθροισμα κρατών μελών. Γιατί ακούμε συχνά ε, τα κράτη να λένε δώστε μας μεγαλύτερη εξουσία για να φροντίσουμε για την ασφάλεια. Ε, δεν είναι αυτή η ελεγγύη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανοντάζα. <clears throat> Ευχαριστώ. Θέλω λίγο να αντιδράσω ε, ε, τα όσα είπατε για την άμυνα, για την εξωτερική πολιτική. Νομίζω ακόμα απέχουμε. Όλα αυτά είναι μάλλον εικασίες σε σχέση με το τι θα κάνει η επόμενη ε, αμερικανική κυβέρνηση και το τονίζω αυτό γιατί δεν αποφασίζει μόνος του και η διοίκηση γενικά. Υπάρχει και το Κογκρέσο και οι Ρεπουμπλικανοί, η πλειοψηφία του δεν ε, σημαίνει η συμπολιτευσιότητα αυτής της απόψης μαζί του. Ε, οι κασίες ε, είναι ακόμα, εντάξει, <laughs> να τρομάζουμε ήδη. Πάντως ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας και συμφωνώ με τα όσα είπατε για την άμυνα τώρα. Συμφωνώ πολύ τους. Τα κείμενα διαδέχονται το ένα το άλλο. Είτε πρόκειται για κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το πρόγραμμα δράσης, είτε για τα κείμενα του Συμβουλίου της κυρίας Μαγκερίνη. Τα περισσότερα αυτά τα έχουμε ξαναδιαβάσει και ποτέ υλοποίησει. Κάθε φορά που βγαίνει η κυρία Μογκερίνη, την είδα και τις προάλλες, πώς το λέμε, με το... Ε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το Στόλτεμπεργκ, και είπε ότι έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Τίποτα συγκεκριμένο δεν υπάρχει. όσοι προθέσεων και αρχών είναι. Ε, δηλαδή, μα δουλεύουν ε, ψιλογαζί κανονικά. Είναι αφόρητο να συνεχίσει κανείς με αυτή την ρητορική υποδιόμενη ότι προχωρούμε ενώ δεν προχωρούμε. Κάθε φορά βάζουμε τη λέξη συγκεκριμένο σε αντικείμενο κείμενο και είμαστε εντάξει. Εσείς πολύ ωραία τα είπατε τεχνικά και διπλωματικά. Το είπε και ο Μίχαελ Γκάλερ. Το επίπεδο φιλοδοξιών που έχει η Ευρώπη. Τι θέλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά τελικά. Ε, στο τέλος όταν συνενώσουμε όλες τις δυνάμεις, ολοκληρώσουμε, κάνουμε κοινέ προμήθειες, κοινό υλικό, κοινέ μονάδες, για να τα κάνουμε τι όλα αυτά. Θα έχουμε το θάρρος κάποια μέρα να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ποιος είναι ο απότερος στόχος. 28 χώρες είναι έτοιμε τελικά να στείλουν στρατεύματα για να πολεμήσουν κάπου στον κόσμο. Στοιχηματίζω ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία ευρωπαϊκή χώρα που να θέλει να το κάνει αυτό ή να είναι πρόθυμη ή να έχουν τα συστήματα λήψη αποφάσεων που να του επιτρέπουν να το κάνουν. Και όλα τα άλλα είναι εικασίε, ότι θέλετε και να δοξάζουμε ένα τον άλλον για τι συνεργασίε Σε τελική ανάλυση, Ποιο είναι ο κοινό στόχος και η κοινή φιλοδοξία, δεν το έχουμε βρει ακόμα, ούτε έχουμε προοδεύσει. Και όταν βλέπω για τις ε, αποστολές που έχουμε της ΕΠΑ ε, και τις επιχειρήσεις, δεν αμφισβητούμε τίποτα. Δεν μας προβληματίζει. Πέντε-έξι χρόνια ε, εκπαιδεύουμε Σομαλούς στρατιώτες. Αποτέλεσμα, το χάος επικρατεί στη Σομαλία. Μεγαλύτερο από ποτέ. Έχουμε να αναρωτηθεί τι κάνουμε εκεί πέρα. Είναι αποτελεσματικό, βοηθάει, όχι. Ε, είμαστε σε ένα hot spot στο Μοκαντήσου και χαιρόμαστε που έχουμε την Ευρωπαϊκή Σημαία. Εκπαιδεύουμε στρατιώτες στο Μαλί. Λείπει ο κύριο Νάρτ, ε, αλλά ε, είναι καλύτερη κατάσταση στο Μαλί. Είμαστε εντάξει, είναι πιο αποτελεσματικό ο στρατό. Καμία σχέση. Μόλι υπάρχει μια μικρή εξέγερση στο βορρά, ε, είναι ε, μια ε, διαδέχεται την άλλη. Έχουμε καμιά εικοσαριά αποστολές, είναι πανάκριβες. Οι άνθρωποι μια χαρά είναι. Εγώ δεν Οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες εκεί επί τόπου που είναι αναπτυγμένα τα στρατεύματα, αλλά ποιος είναι ο στόχος και ποια τα αποτελέσματα. Οπότε, για άλλη μια φορά θεωρώ ότι χάνουμε το στόχο. Επίσης είπατε και εδώ διαφωνώ λίγο μαζί σας, γιατί για τα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως. Λέτε λοιπόν ότι... Ωραία μήπως να φύγουμε από τη λογική της συνεργασίας και να πάμε στη λογική της αμυντικής ολοκλήρωσης. Εντάξει, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε και τον απότερο στόχο, δεν το αποφεύγουμε αυτό. Κατανοώ τη λογική της ολοκλήρωσης ε, για την υποστήριξη, την επιμελητία. Βεβαίως, έχει τη λογική του αυτό, οικονομίε κλίμακας για τις προμήθειε, για την εκπαίδευση, ε, για την ε, βιομηχανική πιστοποίηση, τις δυνατότητες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία και ε, καλό θα ήταν να είναι ολοκληρωμένα και θα βοηθούσε. Για τις λειτουργικές επιχειρησιακές μονάδες, τις μάχημε μονάδες, ποια ολοκλήρωση, με ποιο μοντέλο, με ένα εκτελεστικό αλλά γαλλικό γαλλικό μοντέλο ή κοινοβουλευτικό που ισχύει στη Γερμανία, που χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή. Καλά, ο καθένας έχει την ιστορία του, τις παραδόσεις, τους θεσμούς ε, κτλ. Είδατε τι πρόβλημα έχουμε τώρα με του μάχημους ε, σχηματισμούς, τα battle groups. Ποτέ δεν πρόκειται να το λύσουμε. Δεν πάει να εκφράζουμε ευσεβεί πόθου εδώ στο Κοινοβούλιο να χρησιμοποιηθούν οι μάχημοι σχηματισμοί. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Για ποιο λόγο, γιατί δεν έχουμε του ίδιου κανόνε για ε, την ε, συμμετοχή σε εχθροπραξίες. Δεν λέω ότι θα πρέπει να έχουμε επιθετική πολιτική, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί και τέτοια αποστολή. Είναι τόσο διαφορετικοί οι κανόνες εμπλοκής σε ένα πόλεμο που έχουμε από χώρα σε χώρα και για λόγους πάντα ιστορικούς που δεν πρόκειται να το λύσουμε. Για ποιο λόγο οι Γάλλοι στρατιώτες προτιμούν να φύγουν μόνοι τους να πάει ο Γαλλικός στο, το στο Μαλί. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να είναι πρόθυμη να χάνει άνδρες στο Μαλί, ακόμα και αν πρόκειται για τον εχθρό, τον τζιχαντιστή που απειλεί την Ευρώπη. Ε, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι σίγουρα. Νομίζω ότι δεν ε, προοδεύουμε παρά τα όσα προσπαθούν να μας πουλήσουν Πολύ ωραία επικοινωνία έχει η υπηρεσία εξωτερική δράση. Πολύ ωραία έχουμε ε, το περιτύλιγμα, αλλά το, είναι το περιτύλιγμα δώρου και από μέσα είναι άδειο το δώρο. Δεν έχουμε προχωρήσει από το 2013 για να μην πω ότι έχουμε όπιστο χωρίσει σε σχέση με τις αρχικές φιλοδοξίες μας του 98 και 99. Εγώ διατηρώ πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Παρόλο που χτυπάνε διάφορα καμπανάκια παντού. Η εκλογή του κυρίου Τραμπ για μένα είναι το πιο σοβαρό καμπανάκι, ακόμα πιο πολύ από τον Brexit και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι με 27 δεν πρόκειται να προχωρήσουμε και 26 γιατί η Δανία είναι ήδη έξω. Έχει opt-out. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε κανέναν. Απλώ να είμαστε αρκετά ευέλικτοι έτσι ώστε εκείνοι που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο να προχωρούν περισσότερο. Να του το επιτρέψουν οι άλλοι και όταν είναι έτοιμοι να μπουν και αυτοί. Δεν αποκλείουμε απριόρι κανέναν από χέρι, αλλά να θέλουμε να συμφωνήσουμε για μια παγκόσμια στρατηγική και πώς θα γίνει η άμυνα. Και τελικά ο στρατός ε, σε 27 κράτη-μέλη, χαιρετίσματα. Να ξέρετε, σε 4-5 χρόνια, εγώ δεν ξέρω θα είμαι ακόμα εδώ, να έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας, δεν πρόκειται να έχουμε προχωρήσει ούτε ρούπι και θα εξακολουθούμε να δοξάζουμε ένα τον άλλον για τις αποστολές μας που δεν ανταποκρίνονται στο στόχο, αλλά τις διονίζουμε γιατί έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχουμε στο διεθνές στερεώμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Ναι. Καθηγήτα Μπίσκοπ, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Δυστυχώ δεν μπόρεσα να σα ακούσω γιατί είχαμε ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Ήρθα στο τέλο, ε, έχασα την παρουσίαση, αν και βεβαίω θα με ενημερώσουν οι βοηθοί μου για το τι είπατε. Άρα, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που είπατε. Έχω όμω να σα κάνω κάποιε ερωτήσει. Και θέλω να βασιστώ σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοί μου. Και να σα πω και τη δική μου γνώμη. Δεν πιστεύω ότι η Φεντερίκα πρέπει να πάει στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση. Τίποτα δεν θα απέφερε κάτι τέτοιο. Αντιπαραγωγικό θα ήταν. Ένα τέτοιο ταξίδι. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Η κυβέρνηση δεν έχει σχηματιστεί καν ακόμη. Δεν, δεν, δεν έχουν επιλεγεί όλοι οι υπουργοί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, άλλοι διάβλοι μέσω των οποίων μπορούμε να προσδιορίσουμε τι πρόκειται να συμβεί, ποια είναι τα ενδεχόμενα μπροστά μας. Πιστεύω πραγματικά ότι στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας τα κράτη-μέλη πραγματικά έχουν επιδείξει μια στάση καταστροφική. Οι κυβερνήσεις το ίδιο, η, η ηγεσία μας είναι πραγματικά, ε, πραγματικά καταστροφική. Αυτό ξεκίνησε από την Λέδη ε, Άστον βέβαια, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου, ήταν και ένα βρετανικό ευρύτερα πρόβλημα και τώρα η Φεντερίκα κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί και αξιοποιεί όλες τις περιστάσεις, αλλά χρειάζονται περισσότερα πράγματα και χρειάζεται κάποιον ο οποίος δεν θα θεωρεί ότι είναι απλά ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, αλλά ένα ένας πραγματικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ε, ενεργεί υπέρ της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα θέτει τα κράτη-μέλη ενώπιον των ε, ευθυνών τους. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και λόγω των σχέσεων μας με τη Ρωσία και λόγω της επιθετικής πολιτικής που ασκεί η Ρωσία από την Ουκρανία μέχρι τη Συρία Αλλά βεβαίω, και η κατάσταση με τις ΗΠΑ είναι αυτή που είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή. Κίνα. αναρωτιέμαι. Τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ασφάλειας και της άμυνας, στον τομέα αυτών, έχουν καταβάλει κάποια προσπάθεια να προσδιορίσουν πώς, πόσο έχουμε εγκαταλείψει τον έλεγχο ε, υποδομών στρατηγικής σημασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μιλώ μόνο για τις τεχνολογίες ε, τις αμυντικές τις οποίες έχουμε πουλήσει χωρίς να διατηρούμε κανέναν έλεγχο επί το που καταλήγουν ε, αυτές. Μιλώ για, για υποδομές, μιλώ για βάσεις στρατιωτικές, μιλώ για λιμάνια και, ε, για να μην αναφερθώ καν στις ε, απίστευτες ε, αδυναμίες μας ε, στον κυβερνοχώ, κυβερνοχώρο. Μήπως χρειαζόμαστε ένα Pearl Harbor στον κυβερνοχώρο για να ξυπνήσουμε. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πιέζουμε εδώ και χρόνια για ολοκλήρωση, κοινέ προμήθειες, ανάπτυξη ικανοτήτων, δυνατοτήτων, ε, δεξαμενοποίηση ή τέλο πάντων κοινή χρήση των πόρων. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση και καμία πολιτική ανάληψη δράσης. Γιατί? Δεν είναι οι, οι, ε, ε, ικανότητες που μας λείπουν, ε, ούτε οι δυνατότητες να, να αξιοποιηθούν οι πόροι και ε, οι ικανότητές μας. Ε, αναφέρθηκε και το Μαλί, ε, το οποίο αντικατοπτρίζει πραγματικά μια πολιτική στρατηγική. Άρα ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολες οι περιστάσεις, αλλά όλες οι περιστάσεις είναι δύσκολες. Πάντοτε είναι δύσκολα τα πράγματα. Και παρόλα αυτά κάτι μπορεί να, να επιτευχθεί πάντα η μορφή, και, η μορφή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι πρέπει να γίνει. Μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε αλλαγή ε, σε παγκόσμιο επίπεδο όταν επιτρέπουμε την παράλυση αυτού του, του Συμβουλίου Ασφαλείας από ένα εντελώς παροχημένο σύστημα. δεν ξέρω, ε, ε, ειλικρινά ε, φαντάζομαι, φοβούμε ότι τελικά θα, θα υπάρξει ένα Pearl Harbor στον κυβερνοχώρο μέχρι να ξυπνήσουμε και να αναλάβουμε επιτέλους κάποια σοβαρή δράση. Ευχαριστώ. Ε, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας αυτή και θα ήθελα να σας πω και εγώ τα δικά μου σχόλια και να τα απευθύνω ιδίως στον, στον καθηγητή και βεβαίως στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μπίσκοπ για να μας ε, πει τη γνώμη του για όσα ακούστηκαν. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Συμμερίζομαι και συμφωνώ με τις ε, απόψεις σας ε, όσον αφορά την πυκλομορφία των ε, προκλήσεων, των ερωτηματικών που έχουμε να απαντήσουμε, των διαφορών, των διαιρέσεων, των, ε, της ποικιλία των θέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Να κάνω μία παρατήρηση όσον αφορά την παγκόσμια στρατηγική και τα συμπεράσματα Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013. Πράγματι μοιάζουν τα κείμενα αυτά, αλλά η συζήτηση και το περιεχόμενό της είναι πολύ διαφορετική. Δεν μιλούμε για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αρχίζουμε και μιλούμε όλο ένα και περισσότερο για την ΠΕΣΚΟ, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Μια τεχνικά στοιχεία δηλαδή αυτής της συνεργασίας ή τρόπους με τον οποίο μπορούμε να οθήσουμε αυτούς που δείχνουν μια επιφυλακτικότητα ε, ή εκείνοι που κρατούν ε, πίσω ή έχουν ακόμη και συμφέρον ε, να μην αναλυφθεί η δράση όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο Μάρκ Γιούρεκ, υπάρχουν διάφορα, διάφορες εκδοχές αυτών των προκλήσεων και κάποια κράτη-μέλη κινδυνεύουν περισσότερο από την πολιτική της Ρωσίας, από ό,τι άλλα. Και ως εκ τούτου έχουν ε, συγκεκριμένους ε, στρατιωτικούς, ε, οικονομικούς, διπλωματικούς στόχους σε σχέση με την, με την Ρωσία. Δυστυχώς δεν αναλαμβάνουμε συγκεκριμένη δράση. Φυσικά συζητούμε τις πολιτικές και τη συμπεριφορά της Ρωσίας. Αλλά γιατί ζητούμε περισσότερες ε, διπλωματικές ενέργειες ε, απέναντι στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα ε, συζητούμε τα τυπικά στοιχεία, τα τεχνικά στοιχεία αυτού του πανοράματος ασφάλειας. Δηλαδή ότι η Ρωσία είναι σημαντικός εταίρος και στην Ανατολή και στην ε, Συρία με τις αποτρόπες πράξεις που έχει κάνει η Ρωσία εκεί. Μια ε, θετική ατζέντα ε, θα συμπεριλάμβανε την συμμετοχή όλων σε μια συζήτηση για, την, τον τερματισμό του πολέμου. Και αν τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι θετικά για τον Πούτιν, μπορεί πάντοτε να πιέζει τον Ασάντ για να συνεχίσει την την ε, πολιτική του, κατά του Συριακού λαού και την ε, εξώθηση όλο και περισσότερων ανθρώπων προς την Ευρώπη. Έτσι η, στάση μας θα γίνεται όλο ένα και υπιότερη γιατί στην ουσία εμείς τον βοηθάμε να μας εκβιάζει. Γιατί θέλουμε διπλωματία με τον Τραμπ. Γιατί παρά την κριτική μας η αλήθεια είναι ότι το αίτημα της εκστρατείας του που δεν είναι απαραίτητο ότι θα ε, είναι και ε, πραγματικό αίτημα που θα εκφραστεί και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ε, ούτε είναι σίγουρο ότι είναι και η άποψη των συμβούλων του. Γιατί ήταν αρκετά βολικά αυτά τα αιτήματα που, εκφράστη, που εξέφρασε ο Τραμπ για μεγάλο τμήμα και των ευρωπαϊκών ελίτ Τώρα, θέλουμε να συζητήσουμε ποιος θα υλοποιήσει αυτό το αίτημα ή θέλουμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα παραπέμπουν και στις θεμελιώδεις μας ε, αρχές όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό, την ε, ε, αποτροπή παράνομων προσαρτήσεων ή θέλουμε να κυριαρχήσουν οι οικονομικές αρχές επί της ασφάλειας και του δικαιώματος των, της αυτοδιάθεσης των λαών, τουλάχιστον στην ευρύτερη γειτονιά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Κύριε καθηγητά, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις απόψεις και τα σχόλιά σας όλα. Θα αρχίσω ε, στα αγγλικά, ε, παρόλο που θα μπορούσα να μιλήσω και άλλες γλώσσες, αλλά περνάω τα αγγλικά προς το παρόν. Ο κύριος ε, ρώτησε για τα οικονομικά. Πέντε δισεκατομμύρια είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το χρόνο και πηγαίνετε και αγοράστε ό,τι θέλετε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ε, χρηματοδοτεί την έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θα έρθουν από τα κράτη-μέλη τα ίδια. Δεν τους δίνει χαρτζηλίκι να πάνε να πάρουν όπλα. Και... Ε, είναι καλή ιδέα ε, τα κράτη-μέλη, ε, όμως δεν σπρώχνονται για να υλοποιήσουν την ιδέα αυτή. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο ε, έχει νόημα, ξέρει τι θέλει να το κάνεις. Ε, τώρα έχουμε την ΒΕΣΚΟ, την ε, μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Για τον μηχανισμό ε, Αθηνά Ατένα χρηματοδοτείται από εκεί η ανάπτυξη των μάχημων σχηματισμών, των battle groups. Συμφωνώ με τον κύριο Ταζάν. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν πρόκειται να λύσει το θέμα της μη χρήσης των μάχημων σχηματισμών. Ακόμα και αν έχουμε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του, τι γίνεται με τη χώρα μέλος που ε, μπορεί να το κάνει, ενδιαφέρεται, είναι πρόθυμο. Και για να είμαι σε όλη αυτή την ε, συζήτηση σα συνιστώ να μην αναφέρετε καν τους μάχημου σχηματισμού, γιατί ακόμα και αν το λύσετε αυτό, τι θα έχετε, θα έχετε δύο τάγματα επιφυλακή, ε, που όταν υπάρχει μια κρίση, τι θα σώσουν τα δύο τάγματα ακριβώ, τίποτα. Ε, για τους μάχημους ε, σχηματισμούς χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη ως δικαιολογία για να αποφύγουν τις σημαντικότερες ερωτήσεις και ζητήματα. Τώρα, για το θέμα ε, ε, τον οδηγό του απεσιόδοξου για το 2017 που ρωτήσατε. Για την Κίνα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και η Ευρώπη έχει μια δυσκολία εκεί. Στην τελευταία ε, ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έγινε λόγος για ε, αμοιβαιότητα ε, στις επενδύσεις. Εμείς έχουμε ανοίξει αγορές διάνοιχτα και η Κίνα ερμητικά κλειστή. Οι πολιτείε έχουν πρόβλημα και θεωρούν τον εαυτό τους ε, πρωταθλητή της ελεύθερης ανοιχτής αγοράς, αλλά έχουν και κρίσιμες υποδομές που τις προστατεύουν και γίνεται πολύ σοβαρή συζήτηση γι' αυτό. Και θα πρέπει να είναι πιο εξισορρομένη η συμφωνία με την Κίνα. Ταυτόχρονα όμως να γνωρίζουμε και να διατρανώνουμε ότι ε, δεν θα έχουμε προστατευτισμό σε σχέση με την Κίνα. Ένα άλλο σενάριο που είναι εξίσου επικίνδυνο είναι το εξής Ας φανταστούμε ότι θα υπάρξει και χειρία στη Συρία. προσπαθούμε να εξάγουμε την ευρωπαϊκή ιδέα για τη Μέση Ανατολή, ε, που δεν είναι καλό, είναι οι παγωμένες σειράξει. Θα έχουμε κατάπαυση του πυρό, κρατήδια σταθή και παγωμένα τα πράγματα. Εμείς οι Ευρωπαίοι αυτό θέλουμε, θέλουμε να είμαστε εγγύητρια δύναμη αυτή της κατάπαυση του πυρός, αν όχι. Ε, αυτές οι ομάδες που είναι και χωρίς κράτος, ε, οι αντάρτες, θα ψάξουν άλλο προστάτη. Βλέπετε τη Ρωσία και εκεί θα υπάρχει ε, μια περιοχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει παρουσία και θα είναι και μάλιστα διάφοροι προς εμάς. Και αυτό είναι πιο δύσκολο και θα στραφούν στο Ριάτ, στην Τεχεράνη ή τη Μόσχα αν το κάνουν αυτό αυτές οι αντάρτικες ομάδες και μη χειρότερα. Θα είναι μάλλον αρνητικό αυτό το σενάριο. Αυτό επίσης και με ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω. Ακούσαμε πολλά σχόλια για το μέχρι που θα πρέπει να φτάσουμε ε, στην προσπάθειά μας να συμφωνήσουμε με τη Ρωσία και ποιος συμβιβασμός είναι εφικτός. Τι είδους. Κοιτάξτε, ρεαλιστές θα έλεγα να είμαστε. Προφανώς δεν είναι τέλεια η κατάσταση της μη επιστροφής της Κρυμαίας στην Ουκρανία, αλλά εμεί δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε και δεν μπορούμε να το έχουμε στόχο αυτό. Να σκεφτόμαστε τι είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή να λυθεί η ε, σύραξη στην Ανατολική Ουκρανία, στον Τον Γιατί ούτε και έχουμε συμφέρον να διατηρηθεί μια παγωμένη σύραξη στην παγκόσμια στρατηγική κάπως παίρνουμε αποστάσεις από τον εκδημοκρατισμό. Δεν μπορείς να εκδημοκρατήσεις μια χώρα έξωθεν. Αν θέλει να εκδημοκρατιστεί μια χώρα, μπορείς να την υποστηρίξεις, αλλά δεν μπορείς να εξάγεις εκδημοκρατισμό. Δεν μπορείς να το εφεύρεις έτσι, μια μηχανική εμφύτευση δημοκρατίας. Το ξέρω ότι μπορεί να μας αρέσει, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι γίνεται με τις δικές μας ε, δημοκρατίες. Ε, ε, απελούνται, απειλείται η Ευρώπη από το εξωτερικό όπως είναι στην Ουκρανία ή από το εσωτερικό όπως είναι στην Τουρκία. Αυτό είναι μεγαλύτερο θέμα. Ακόμα και αν λέμε ότι δεν μπορούμε να εκδημοκρατήσουμε μη δημοκρατικά καθεστώτα, μπορούμε να παίξουμε ρόλο ως εγγυητής της δημοκρατίας εκεί που ήδη υπάρχει στη γειτονιά μας και απειλείται. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει και αυτό να απαντηθεί. Έχει δίκιο ο κύριος Δόζο ότι τελικά είναι λίγα τα κράτη-μέλη εκείνοι που είναι πρόθυμα να μπουν στο πραγματικό πόλεμο όταν χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι ε, ε, επεμβατιστής, αλλά δεν μπορείς να είσαι και ειρηνιστής όταν θέλεις να υπερασπιστείς κάποιες αξίες. Όταν είσαι ειρηνιστής κάποιες φορές σηκώνεις τα χέρια ψηλά και εντάξει. Και απεμπολίσει και τις αξίες σου. Επειδή λοιπόν είναι λίγα τα κρατημέλη που έχουν τη βούληση να μπουν σε πόλεμο όταν αυτό είναι αναπόφευκτο, ε, μάλλον όταν ε, χρειάζονται επιχειρήσεις αυτές θα είναι ad hoc κάθε φορά, μεμονωμένε. Βλέπουμε για τη Γαλλία ο πρώτος εταίρος στα στρατιωτικά θέματα παραμένει ο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Θα βγει από την ΕΠΑ όμως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία δεν θα στραφεί αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ. Μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Και όταν στείλουν ε, τέτοιες, ε, ε, τέτοιες επιχειρήσεις το κάνουν εκτός των δομών και του ΝΑΤΟ και τα, θα συνεχίσουν να το κάνουν όπως μέχρι τώρα και δεν είναι πάρα πολύ θετικές όλες αυτές οι προοπτικές. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να θέσω. Η Άννα Γκόμες έχει δίκιο. Να μην πάει τώρα στον Τραμπ η Μοκερίνη, τι να κάνει, τουλάχιστον πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Είδαμε τι έπαθε ο Άμπε και πώς η κοινή γνώμη της Ιαπωνίας το θεώρησε μάλλον ταπείνωση. Τον δέχτηκαν ο Ντόναλτ και η Βάνκα, κοντζάν πρωθυπουργό. Και καλύτερα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυρία Μογκερίνη το χρόνο ε, να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, μια ε, ε, πρόταση και αυτή τη στιγμή αναλάβει να πάμε και να πούμε ειδού τι θέλουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ε, ή να πούμε κάτι για τον Άτο. πια πράγματα που είναι τελείως στον αέρα ακόμα. Αυτά. Σταματώ εδώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάλι για τα σχόλιά σας. Καθηγητά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα ενώπιό μας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές και τους υπολείπους συμμετέχοντες. Τα επόμενα δύο σημεία στη μέση διάταξη θα συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών. θα παρακαλούσα να αποχαιρετήσουμε ε, ε, των προσκεκλημένων μας και επιτρέπεται να παρευρίσκονται μόνο ε, ευρωβουλευτές και πολιτικοί σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που δικαιούνται να ε, παρευρίσκονται. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλούν